No, no, no, no. It was in, um, Ας ξεκινήσουμε λοιπόν. Συνεχίζουμε ουσιαστικά την συζήτηση που ξεκινήσαμε με τον Υπουργό Εξωτερικών της Αλβανίας σήμερα το πρωί έχουμε ε, μια πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τη διαδικασία ένταξης Αλβανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα ζητήσω λοιπόν από τον κύριο Χουντή, ο οποίος είναι ο εισηγητής, να πάρει το λόγο και να μας κάνει μια σύντομη παρουσίαση. Μια σύντομη παρουσίαση των προτάσεών του. Κύριε Χουντή, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ζητώ συγγνώμη για αυτή την καθυστέρηση. Η υποχρέωσή μου σε μια άλλη επιτροπή και η εντύπωση ότι το θέμα είναι αργότερα ε, μου δημιούργησε αυτή την καθυστέρηση. Ζητώ και πάλι συγγνώμη. Πείτε μου σας παρακαλώ κύριε Πρόεδρε πόσο χρόνο έχω στη διάθεσή μου για την παρουσίαση της έκθεσης. Uh, uh, Εφτά λεπτά 5 λεπτά, 7 λεπτά, αυτό θα σας έλεγα πάνω κάτω. Είμαι αρκετά γενναιόδωρος. Ευχαριστώ και πάλι. Ε, θέλω να σημειώσω το γεγονός ότι η συζήτηση της έκθεσης για την ενταξιακή προοπτική της Αλβανίας σήμερα στην Επιτροπή μας συνδυάζεται από το γεγονός ότι στην πρωινή συνεδρίαση είχαμε μια επίκαιρη συζήτηση για την κατάσταση στην Αλβανία και τα προβλήματα με τον Αντιπρόεδρο της Αλβανικής Κυβέρνησης και Υπουργό Εξωτερικών και κατά συνέπεια είχε τη δυνατότητα η Επιτροπή, ε, αρκετοί συνάδελφοι που είμαστε παρόντες και παρούσες στην πρωινή συνεδρίαση, να ρωτήσουν, να εκφέρουν γνώμη σχετικά με την κατάσταση στην Αλβανία. Ε, το κείμενο το έχετε μπροστά σας και προφανώς περιμένω με ενδιαφέρον και με ανοιχτή διάθεση της παρατηρήσης των συναδέλφων. Ε, έχω την εντύπωση πως τα βασικά υπάρχει συμφωνία στις διαπιστώσεις και στις επισημάνσεις, αλλά οι παρατηρήσεις που θα γίνουν θα βοηθήσουν στη βελτίωση του κειμένου. Θέλω από την αρχή να ευχαριστήσω ε, όσους βοήθησαν για τη σύνταξη της έκθεσης, ιδιαίτερα τη γραμματεία της ΑΦΕΤ, την ΕΒΑ. Ε, για τη σύνταξη του κειμένου είχα συνεργασία με την αντίστοιχη επιτροπή της Κομισιόν η συνεργασία μου με την ε, αλβανική πρεσβεία ήταν συστηματική, ε, όμως την επικαιροποίηση των στοιχείων και, τη και τις διαπιστώσεις με βοήθησε η πρόσφατη επίσκεψη που έκανα στην Αλβανία, όπου συναντήθηκα με την πολιτιακή και πολιτική ηγεσία, με όλα τα κοινοβουλευτικά πολιτικά κόμματα, υπογραμμίζω με όλα τα κοινοβουλευτικά πολιτικά κόμματα, όχι μόνο με την κυβερνητικό κόμμα και το αντιπολιτευόμενο, αλλά με όλα τα, ε, τα κοινοβουλευτικά κόμματα, με σημαντικά με υπουργού που κατέχουν σημαντικό χαρτοφυλάκιο και που άπτονται των θεμάτων που μας αφορούν και επίσης υπογραμμίζω το γεγονός ότι ε, συναντήθηκα με εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών, δηλαδή με εκπροσώπους συνδικάτων, με συλλόγους που αγωνίζονται κατά της εμπορίας παιδιών, με την Ένωση Αλβανών Δημοσιογράφων, με την οργάνωση Ρωμά Active Albania, με γυναί... Ε, οργανώσεις που υποστηρίζουν τα δικαιώματα των γυναικών. Το θεωρώ σημαντικό, με βοήθησε πολύ, διότι ε, η εικόνα που υπάρχει και τα προβλήματα βιώνονται από μια ατροφική κατά τα άλλα κοινωνία των πολιτών. Ε, γενικά, στην έκθεσή μας νομίζω ότι πρέπει να επιβεβαιώσουμε την πρόθεση του Κοινοβουλίου ε, για να υποβοηθήσει και να υποστηρίξει την ένταξη όλων των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θεωρώντας ότι αυτό, αυτό μπορεί να αποτελέσει και κίνητρο για εντατικοποίηση των προσπαθειών, αλλά και ταυτόχρονα αυτή η διαδικασία μπορεί να βοηθήσει την αλβανική κυβέρνηση και τις αλβανικές πολιτικές δυνάμεις και κοινωνικές δυνάμεις να αντιμετωπίσουν προβλήματα που έχουν να κάνουν με τον εκδημοκρατισμό, και με τη βελτίωση του βιωτικού επίπεδου των πολιτών. Επίση, η αντιμετώπιση των προβλημάτων, αναφέρομαι σε γενικέ παρατηρήσει, ορισμένων τουλάχιστον, βοηθούν επί τη ουσία την καλή γειτονία με άλλε χώρε, μια και η αντιμετώπιση του δεν αφορά μόνο την Αλβανία, α πούμε τα φαινόμενα τη διαφθορά, τα φαινόμενα τη ε, διακίνηση μαύρου χρήματο, τα φαινόμενα του τράφικινγκ, αν δεν συμβάλλουν όλε οι γειτονικέ χώρε, πέρα από τι προσπάθειε τη αλβανική πολιτεία, δεν θα μπορέσει να αντιμετωπιστεί. Να αντιμετωπιστούν. Κατόπιν τούτου η αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων προφανώς βοηθούν τη σταθερότητα και τη συνεργασία των χωρών της ε, περιοχής. Και τέλος, σε, σε αρκετά σημεία, σε ορισμένα σημεία, η διατύπωση του προβλήματος έχει το χαρακτήρα ότι οφείλουμε ω Ευρωπαϊκή Ένωση και ω Ευρωπαϊκό ε, Κοινοβούλιο να βοηθήσουμε με ε, πακέτα χρηματοδότησης με τεχνογνωσία στην αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων. Το πρώτο πρόβλημα, μπαίνοντα πιο αναλυτικά, είναι αυτό που συζητήθηκε εκτενώς και που απασχολεί όλους. Είναι η κατάσταση που έχει προκύψει στην ε, Αλβανία μετά τις πρόσφατες, πρόσφατες εν πάση περιπτώσει, εκλογές του προηγούμενου Ιουνίου. Έχει δημιουργηθεί ένα αδιέξοδο. Το αδιέξοδο αυτό δεν φαίνεται να λύνεται εμφανίζεται ως σύγκρουση ε, της κυβέρνησης και της αντιπολίτευσης σχετικά με την εγκυρότητα του αποτελέσματος των εκλογών δεν φαίνεται διέξοδος από αυτή τη λύση. Κατά την άποψή μου και κατά την εικόνα που αποκόμισα, εκφράζονται παθολογίες ενός πολιτικού συστήματος που χρειάζεται βαθιά βήματα εκδημοκρατισμού. Σε κάθε περίπτωση αυτό το αδιέξοδο το πολιτικό δεν επιτρέπει να αντιμετωπιστούν άλλες πολιτικές και θεσμικές δυσλειτουργίες και δυσκολεύει εξ αντικειμένου, θα έλεγε κανείς, και τις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις ή τα βήματα που πρέπει να γίνουν σε αυτή την περίοδο. Εδώ υπάρχει μια συζήτηση και οφείλω να την πω ανοιχτά τι μπορεί να κάνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Επιτροπή μας, τι μπορεί να κάνουν οι ευρωπαϊκοί θεσμοί. Η, άποψη ότι πρέπει εμείς να υποδείξουμε δεν με βρίσκει σύμφωνα. Μια τέτοια υπόδειξη μάλλον δεν θα γίνει αποδεκτή από το σύνολο του, του πολιτικού κόσμου της Αλβανίας, ο οποίος πρέπει να λύσει το πρόβλημα, ενώ ταυτόχρονα κάθε δήλωση τέτοια ή άλλα, η άλλη η διαφορετική, αξιοποιείται μέσα στην πολιτική διαμάχη που είναι οξύτατη στην περίπτωση, στην, ε, αυτή την περίοδο. Επομένως, να προτρέψουμε να βρεθεί λύση η διαφορετικη αξιοποιειται μεσα στην πολιτικη διαμαχη που ειναι οξυτατη στην στην αυτη την περιοδο επομενως να βγάζει από αυτό το αδιέξοδο, να μπορέσει να λειτουργήσει σε να... υπάρξει πλήρης λειτουργία της... του Κοινοβουλίου και εξασφάλιση του πολιτικού πλουραλισμού καθώς ε, τον επόμενο χρόνο θα υπάρχουν τοπικές εκλογές. Αυτή η καχυποψία, αυτή η ανα... αβεβαιότητα, αυτά τα αδιέξοδα προφανώς δεν θα βοηθήσουν και την κανονική τυπική δημοκρατική διαδικασία των εκλογών, επαναλαμβάνω, της επόμενης περίοδου. Επειδή ο χρόνος είναι περιορισμένος, θα κωδικοποιούσα τις παρατηρήσεις μου σε τρία, αν μου επιτρέπετε, σημεία, τρεις μεγάλες, ε, τρία μεγάλα θέματα, τρεις μεγάλες κατηγορίες. Ε, το πρώτο, τρία μεγάλα θέματα. Το πρώτο είναι το θέμα των θεωρήσεων. Νομίζω ότι πρέπει να υποστηρίξουμε ότι ε, την απελευθέρωση της βίζας αυτό κάνει η έκθεση και η Επιτροπή πρέπει με καινούργια πρόταση να το όσο γίνεται πιο γρήγορα αυτό το θέμα. Θα ήθελα όμως να σας ε, εξομολογηθώ στο πλαίσιο της Επιτροπής ότι στο πλαίσιο μιας τέτοιας θέσης, υποστήριξης πραγματικά της απελευθέρωσης, δεν πρέπει να παραβλέπουμε δύο σημεία. Ε, το ένα είναι τι θα συμβεί αν υπάρξει αυτή η απελευθέρωση όσο αφορά μετακίνηση ενδεχομένως μαζική Αλβανών πολιτών προς το εξωτερικό και το δεύτερο σε κάθε περίπτωση επειδή η τεχνική προετοιμασία έτσι κι αλλιώς έχει γίνει έτσι κι αλλιώς έχει γίνει, υπάρχει ένα θέμα όλα αυτά τα προσωπικά δεδομένα που συγκεντρώνονται, ποιος τα ελέγχει, ποιος τα διαχειρίζεται και αν υπάρχει η προστασία των προσωπικών δεδομένων. Η δεύτερη κατηγορία των παρατηρήσεών μου έχει να κάνει γενικά με το χώρο των θεσμών και των δικαιωμάτων, του νομοθετικού πλαισίου. Εδώ πράγματι έχουν γίνει βήματα νομοθετικά, σωστοί νόμοι έχουν ψηφιστεί. Το κεντρικό πρόβλημα είναι η εφαρμογή του στην πράξη. Και εδώ είναι η παρατήρηση που είπα στην αρχή, ποια θα είναι η βοήθεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ε, αν χρειαστεί σε συγκεκριμένα θέματα να σας πω ακριβώς τι εννοώ επ' αυτού, ούτω ώστε αυτέ οι προσπάθειε να έχουν πρακτική εφαρμογή. Και η τρίτη και τελευταία παρατήρηση, γιατί ξέρω ότι εξάντλησα τον χρόνο, έχει να κάνει με τα ζητήματα τη οικονομία. Σε ποια οικονομική κατάσταση βρίσκεται η Αλβανία. Ομολογώ, όπω και σε άλλα σημεία που ενδεχομένω στην πορεία τη συζήτηση ε, αναφερθώ για την ενημέρωση των συναδέλφων ότι χρειάζεται μια επικαιροποίηση. Η διαπίστωση που γράφεται μέσα στην έκθεση ενδεχομένως είναι σκληρή από τη δική μου την πλευρά, όμως πρέπει να αναγνωριστεί ότι πράγματι η Αλβανία και το τελευταίο διάστημα μέσα σε συνθήκες κρίσης είχε υψηλού ρυθμούς ανάπτυξης, οι ενστάσεις και τα ερωτηματικά είναι αν αυτή η ανάπτυξη είναι, ε, βασίζεται πάνω σε πραγματικά δεδομένα, καθώς υπάρχουν ανησυχητικά σημάδια στον ορίζοντα, δηλαδή μεγάλο μέρος της οικονομίας της Αλβανίας στηρίζεται στα εμβάσματα και στις επενδύσεις Ελλάδας, Ιταλίας τουλάχιστον και επειδή αυτές οι χώρες είναι σε κρίση, δεν ξέρω αν αυτό η ροή συνεχιστεί, επομένως είναι ένας παράγοντας αμφίβολος. Το δεύτερο είναι ότι στηρίζει πολλά στον κατασκευαστικό τομέα όπου έχουμε μείωση και το τρίτο είναι, με βάση στοιχεία του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, υπάρχει μείωση των ιδιωτικών επενδύσεων. Αυτό το ερωτηματικό σχετικά με το ότι θα έχουμε την κρίση ίσως καθυστερημένα δεν πρέπει να μα μας κάνει και εγώ είμαι έτοιμος να το διορθώσω ότι εν πάση περιπτώσει υπάρχει μια ανάπτυξη του 3% να τη γίνει βιώσιμη με μια σειρά άλλα μέτρα. Ε, επειδή καταλαβαίνω ότι το θέμα, ε, ο χρόνος έχει περάσει, λέω κάτι που υπόθηκε ε, κατά την πρωινή συζήτηση που έχει να κάνει με το ενεργειακό και την προστασία του περιβάλλοντος και τελειώνω με αυτό. Σε σχέση με το ενεργειακό, σαφώς πρέπει να γίνουν, επειδή ξεκινάει αυτή η ανασυγκρότηση, ας το πούμε, η ενεργειακή εξασφάλιση, από την αρχή πρέπει να υπάρχει προτεραιότητα στις ανανεώσιμες πηγές ε, ενέργειας. Το δεύτερο πρέπει να γίνει συνεργασία με τις γειτονικές χώρες, καθώς όλα αυτά τα θέματα αφορούν και τις γειτονικές χώρες και το μελλοντικό στάτους σχέσεων. Αναφέρω αυτό που ανέφερε η συνάδελφος Κοπά το πρωί για την πιθανότητα δημιουργία πυρηνικού εργοστασίου κοντά στα ελληνικά σύνορα και γενικότερα ένα πρόβλημα που υπάρχει ε, σχετικά με την αν η πυρηνική ενέργεια, ε, κατά την άποψή μου όχι, αποτελεί ε, εναλλακτική μορφή ενέργειας. αυτά με συγχωρείτε και πάλι για την καθυστέρηση, με συγχωρείτε αν τράβηξε παραπάνω η εισήγηση. Περιμένω τις παρατηρήσεις με ενδιαφέρον και να δούμε μετά με ποιον τρόπο να θα δουλέψουμε, ούτω ώστε να έχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για την Επιτροπή. Σα ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, ο κύριος Κούκαν, που είναι πρόεδρος της αντιπροσωπείας. Παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Είμαι σαφώς υπέρ της έκθεσης αυτής και θεωρώ ότι μπορεί να αποτελέσει σημείο κίνησης για περαιτέρω συζητήσεις. Θα ήθελα να τονίσω κάποια ζητήματα, κάποια πολιτικά ζητήματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σαφώς όλοι γνωρίζουμε ότι υπάρχει ένα πρόγραμμα ομαλοποίησης της πολιτικής κατάστασης στην Αλβανία. Πρέπει λοιπόν να τονίσουμε το ζήτημα αυτό, ιδίως στα πλαίσια των μελλοντικών ευρωπαϊκών φιλοδοξιών των Αλβανών. Είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι η λύση στην κατάσταση θα πρέπει να βρεθεί μέσω των δημοκρατικών θεσμών και ότι όλες οι πολιτικές ομάδες θα πρέπει να δεχθούν τα αποτελέσματα. Επίσης θεωρώ ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να λάβει θέση επί του ζητήματος και αν κρυθεί αναγκαίο θα πρέπει να κάνει οτιδήποτε μπορεί προκειμένου να βοηθήσει την κατάσταση προς την ομαλοποίησή της. Ο κύριος συγητής θα πρέπει ίσως να αναφέρει στην εκθεσή του ότι η Αλβανία υπέβαλε το, τις απαντήσεις στο πλήρες ερωτηματολόγιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Προφανώς ο συγητής δεν το γνώριζε αυτό τη στιγμή της σύνταξης της ε, έκθεσης. Νομίζω ότι θα πρέπει να συμπληρώσουμε απλώς την έκθεση και με το στοιχείο αυτό, ότι έχουν πια δοθεί απαντήσεις. Θα ήθελα επίση να ενθαρρύνω τον ε, εισηγητή, όπω είπε και αυτό, να τροποποιηθούν οι παράγραφοι αυτοί που έχουν να κάνουν με την οικονομική κατάσταση στην Αλβανία, 22 με 25 τις παραγράφους αυτές, γιατί όσοι έχουν αυτή τη στιγμή νομίζω ότι απέχουν κάπως από την πραγματικότητα. Δεδομένου το ότι η Αλβανία είναι μια φτωχή χώρα και το ότι κατάφερε τελικά να αντισταθεί σχετικά καλά στην οικονομική κρίση, ακόμα και συγκρινόμενη με άλλες χώρες της ε, περιοχής. Αυτό είναι θετικό. Η θετική αύξηση του ΑΕΠ πέρυσι, για παράδειγμα, Νομίζω λοιπόν ότι θα πρέπει να αντικατοπτρίζεται εδώ πέρα η πραγματικότητα λίγο πιο αντικειμενικά και επομένως οι παράγραφοι αυτοί θα πρέπει να τροποποιηθούν. Επίσης θα πρέπει να αφαιρθούμε στον ενεργό ρόλο που διδραματίζει η Αλβανία στα πλαίσια της περιφερειακής συνεργασίας στα Βαλκάνια. Νομίζω ότι επίσης θα πρέπει να αναφερθεί ότι έχει καταργήσει τις απαιτήσει θεωρήσεων για άλλες χώρες στην περιοχή, για τη Σερβία για παράδειγμα, και νομίζω ότι θα πρέπει να γίνεται ένα σχόλιο σε σχέση με αυτό. Προφανώς υπάρχουν ε, ακόμα πολλά ζητήματα που εκκρεμούν για την Αλβανία, για τα οποία η Αλβανία θα πρέπει να εργαστεί σκληρά, προκειμένου να προωθηθεί περισσότερο η πορεία της προς την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Ωστόσο, θεωρώ ότι ε, η έκθεση αυτή θα πρέπει να ενθαρρύνει θετικά την ε, Αλβανία χωρίς να αποκρύπτει τίποτα έτσι ώστε να μπορούμε και να επικρίνουμε αντικειμενικά, αλλά να μπορούμε παράλληλα να φερόμαστε και στα θετικά επιτεύγματα της χώρας. Συμφωνώ με τον εισηγητή όταν λέει ότι το καθεστώς απελευθέρωσης των, στα πλαίσια της ελευθέρωσης των θεωρήσεων είδαμε σημαντική πρόοδο και ότι θα πρέπει να ενθαρρύνουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υποβάλει τις απαραίτητες προτάσεις σύντομα προκειμένου να καταφέρουμε να αναλάβουμε δράση γρήγορα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Νομίζω λοιπόν ότι με τις τροποποιήσεις αυτές θα καταφέρουμε να έχουμε μια αντικειμενική αξιολόγηση της Αλβανίας. Το λόγο έχει η κυρία Πακ. Ναι, Ευχαριστώ πολύ τον εισηγητή, αλλά πρέπει να πω ότι η έκθεση αυτή, σε αντίθεση με την τελευταία έκθεση για την Αλβανία, του συναδέλφου Ρούτσεκ, είναι αρκετά αρνητική. Παρόλο που στο μεταξύ έχουν γίνει πράγματα για τα οποία τσακωνόμαστε 10 χρόνια. Δεν νομίζω ότι μπορούμε έτσι με κάποια ε, ελαφρότητα, χαλαρότητα, ελαφρά την καρδία να πούμε εντάξει, καλή έκθεση. Ε, στο παρελθόν έχουμε, στήσει, έχουμε στείλει συγγνώμη, πολύ πιο θετικά μηνύματα και λυπάμαι που ε, δεν ε, βγαίνουν πιο έντονα αυτά τα θετικά. Ε, μιλάτε για το πολιτικό σύστημα, ότι βελτιώνεται. Δεν θα συνεισφέρουμε όμως αν τα αποσιωπήσουμε όλα. Νομίζω ότι είναι δικό μας καθήκον ε, και αποστολή να απευθυνθούμε σήμερα στην αντιπολίτευση όπως κάναμε και στους άλλους στο παρελθόν ότι οι διαμαρτυρίες στους δρόμους και ε, η μη συνεργασία στο Κοινοβούλιο δεν είναι τρόπος να ε, ε, κυβερνάει κανείς ένα δημοκρατικό κράτος και να το λέμε με το όνομά του. Και εγώ περιμένω από μια αντιπολίτευση να τα λέει αυτά στο Κοινοβούλιο. Γι' αυτό την έχουν εκλέξει, όχι για να βγαίνει στους δρόμους. Να τα λέει και το κείμενο. Και όχι να κινηθούν οι πάντες να ζητάμε. Ναι, να κινηθούν, αλλά να πάνε στη Βουλή και να συζητάνε. Και αυτά που δεν μπορεί κανείς να τα λύσει στο Κοινοβούλιο, και πρέπει να πάει στο δικαστήριο, στην εφορευτική επιτροπή, να λυθούν εκεί, εκεί που ορμοζει να ε, προσφύγουν. Ε, παρακαλώ αγαπητέ συνάδελφοι, το σημείο 4 πραγματικά ε, υπερβάλλει. Η έκθεση Ντύρ είναι σαφής. Δεν μπορείτε να βγαίνετε και να ε, μιλάτε για εκφοβισμό και άσκηση πίεσης και τα λοιπά. το ΟΝΤΙΡ νομίζω είναι σαφές να μην μπούμε σε λεπτομέρειες τέτοιες, γιατί ούτε εσείς, ούτε εγώ παρόλο που ήμουν παρούσα, έχουμε άποψη γι' αυτό. Και για τα οικονομικά θα πρέπει να είμαστε λίγο πιο προσεκτικοί. Εξηγήστε μου, τι σημαίνει το άρθρο 23. Θεωρεί ότι η Αλβανία θα πρέπει να επιλέξει τι δέουσε οικονομικέ πολιτικέ που θα εξασφαλίσουν βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη. Ωραία, και τι λέει αυτό το πράγμα. Τίποτα. Ποια μέτρα δεν έχει αρκετή ουσία για μένα το θέμα αυτό και ξαφνικά στο 24 γίνεται λόγος για την παιδεία. Λες και είναι όλα στραβά και στην παιδεία. Τότε παραμελούμε και ξεχνάμε αυτά που γίνανε στην παιδεία τα τελευταία χρόνια. Την τελευταία δεκαετία έχουν γίνει τεράστιες πρόοδοι στην παιδεία. Παρακαλώ ε, να ξεχωρίζουμε ε, τις διάφορους τομείς πολιτικής με κάποια προσοχή και επιμέλεια. Α, θα κάνω τροπολογία τώρα. Ε, δικιά μου, θα σας παρακαλούσα τώρα να μην αρχίζετε πάντα με τα αρνητικά τη παραγράφου σα. Μπορείτε να αρχίσετε και με θετικό καμιά φορά, και, αλλά το τάδε πρέπει να βελτιωθεί. Είναι και πιο χρήσιμο ε, για να γίνει και αποδεκτή η έκθεση. Τα είπα αρκετά γρήγορα, λέει η κυρία Πακ, βεβαίω, Ο κύριος Ρότσεκ. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, θα είμαι και εγώ σύντομο. Να ευχαριστήσω τον κύριο Χουντή για την πολύ καλή εργασία του. Διάβασα πολύ προσεκτικά την ε, έκθεση. Θεωρώ ότι ε, Μπορεί να είναι μια πολύ καλή έκθεση, αλλά όπως είπε και η συναδελφός μου θα πρέπει να γίνουν κάποιες βελτιώσεις. Συμφωνώ με την ε, Doris ε, Πακ ότι είναι πολύ σημαντικό να ενθαρρύνουμε τις μεταρρυθμίσεις. Όχι μόνο τους επισήμους, τους πολιτικούς, αλλά και τους ίδιους τους, πολιτικούς, τους πολίτες, με συγχωρείτε, να ενθαρρύνουμε. Ενδεχομένως, λοιπόν, θα μπορούσαμε να υιοθετήσουμε μία προσέγγιση όπου θα ξεκινάμε με τα θετικά, με τα επιτεύγματα, τα τελευταία δύο-τρία χρόνια έχουν γίνει πολλά επιτεύγματα, έχει επιτελεστεί πρόοδος και σαφώς στη συνέχεια μπορούμε να εντοπίσουμε και τα προβλήματα. Ακόμα και δούμε την πολιτική κατάσταση, την παράγραφο 3 για παράδειγμα. Ναι, όντως υπάρχει μια πολιτική κρίση. Αλλά δεν μπορούμε να μιλάμε για θεσμική κρίση, γιατί μόλον ότι υπάρχει μποϊκοτάρισμα από την αντιπολίτευση στο Κοινοβούλιο, το Κοινοβούλιο λειτουργεί και έχουν περάσει γύρω στους 150 νόμους, για παράδειγμα. Πολύ περισσότερους δηλαδή από ό,τι στην προηγούμενη θητεία του Κοινοβουλίου. Νομίζω λοιπόν θα πρέπει να το λάβουμε αυτό υπόψη μας. Όσον αφορά την πολιτική κατάσταση, ναι, το είπα και σήμερα το πρωί, πρέπει να μείνουμε στις αρχές. Στα πλαίσια μιας κοινοβουλευτικής δημοκρατίας η καρδιά του συστήματος είναι το κοινοβούλιο. Είτε μας αρέσει είτε όχι το αποτέλεσμα των εκλογών, όλες οι πολιτικές ομάδες θα πρέπει να το δεχτούν. Αν υπάρχουν διαφωνίες, αν υπάρχει αίσθημα αδικίας, τότε τα πολιτικά κόμματα θα πρέπει να επιλύσουν το ζήτημα αυτό, θα πρέπει να συζητήσουν, θα πρέπει να κάνουν προτάσεις, θα πρέπει να θεσπίσουν επιτροπές, αλλά στα πλαίσια του Κοινοβουλίου. Ο εισηγητής μας μας είπε ότι κοιτάει λίγο το νομικό πλαίσιο, δεν κοιτάει μόνο τους νόμους που έχουν εγκριθεί και τους θεσμούς, αλλά πώς εφαρμόζονται οι νόμοι αυτοί στην πράξη. Αυτό είναι πολύ καλό, πολύ θετικό, πολύ υγιής η προσέγγιση αυτή. Δεν θα εξετάσω τώρα την έκθεση άρθρο προς άρθρο, γιατί αυτό θα πετούσε πάρα πολύ χρόνο. Ήδη το είπα σήμερα το πρωί και έθεσα κάποιες ερωτήσεις σε σχέση με αυτό. Αναφέρομαι στην οικονομική κατάσταση στην οικονομική ανάπτυξη. Νομίζω ότι οι παράγραφοι αυτές 22, 23, 24 θα πρέπει να λένε κάπου τουλάχιστον ότι η Αλβανία με την Πολωνία ήταν από τις λίγες χώρες που γνώρισαν οικονομική ανάπτυξη και θα πρέπει κάπου να λέμε ότι ε, η χώρα χρειάζεται αυτή την ε, βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη. Νομίζω ότι θα μπορούσαμε μέσω τροπολογιών να το διευθετήσουμε αυτό. Αναφερθήκαμε επίσης στην περιφερειακή συνεργασία και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Θα πρέπει και εδώ όμω να γνωρίσουμε το θετικό ρόλο που διαδραματίζει η χώρα στην περιφέρεια των Βαλκανίων. Η Αλβανία συμπεριφέρεται με ένα πολύ υπεύθυνο τρόπο και νομίζω ότι θα πρέπει να το αναγνωρίσουμε αυτό και θα πρέπει να ενθαρρύνουμε την χώρα να συνεχίσει να διαδραματίζει το ρόλο αυτό και στο μέλλον. Δηλαδή, να ενδυναμωθεί η περιφερειακή συνεργασία και να περάσει μέσω από την οικονομική συνεργασία. Αν δούμε τα στατιστικά δεδομένα που έχουμε στα χέρια μας αυτή τη στιγμή, βλέπουμε ότι οι οικονομικές συναλλαγές, οι εμπορικές συναλλαγές ανάμεσα στις χώρες της περιοχής είναι ακόμα πολύ περιορισμένες. Τώρα το ζήτημα της πυρηνικής ενέργειας και αυτό αναφέρεται. Είναι πολύ νωρίς πιστεύω τώρα να συζητάμε για το ζήτημα αυτό. Δεν έχει λάβει κάποια απόφαση η Αλβανία όσον αφορά την πυρηνική ενέργεια. Δεν μπορούμε λοιπόν να εμποδίσουμε τη χώρα αυτή να πτήσει μορφές ενέργειας, ακόμα και αν πρόκειται για την πυρηνική ενέργεια. Εδώ δεν το κάνουμε αυτό για τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν έχουμε το δικαίωμα να ζητήσουμε από μια χώρα που δεν είναι καν μέλος της Ένωσης, στη φάση αυτή τουλάχιστον, να αναπτύξει ή να μην αναπτύξει συγκεκριμένες ενεργειακές πολιτικές. Θα υποβάλουμε λοιπόν σχετικές τροπολογίες. Ευχαριστώ. 5 Μαΐου 12 το μεσημέρι είναι η προθεσμία υποβολής τροπολογιών. Κυρία Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εχθές, στην Επιτροπή Δημοσίων Ελευθεριών, ε, όπου είμαι σκιώδης εισηγήτρια εγώ για την απελευθέρωση της θεώρησης για την Αλβανία και τη Βοσνία, συζητήσαμε τις πρόοδους που έχει κάνει η Αλβανία Σήμερα το πρωί είχαμε τον Υπουργό Εξωτερικών. Την περασμένη εβδομάδα, την προπερασμένη, είχαμε τον Υπουργό Εσωτερικών ε, που μας επισκέφθηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και ακούγοντάς τους, έχω την εξή εντύπωση. Ο εισηγητή μα έχει κάνει πολύ καλή έκθεση που σίγουρα θα βελτιωθεί και με τι τροπολογίε. Δεν είναι υπερβολικά σκληρό. Όχι είπατε ότι φοβάστε με πως θα λέτε πολύ σκληρά. Όχι. Ακούγοντας τους υπουργούς της Αλβανίας, Θέλουν και αυτοί να έχουν ένα σαφέ μήνυμα, να ξέρουν πού πηγαίνουν, τι πρέπει να κάνουν. Πρώτον, απελευθέρωση τη θεώρησης διαβατηρίων. Αν κατάλαβα καλά, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα αρχίσει να κάνει κάποιες κινήσεις έτσι ώστε το Σεπτέμβριο να ε, φτάσουμε βέβαια πάντα ε, ακούγοντας και τι έχουμε να πούμε εμείς και το Συμβούλιο. Και μελλοντικά ε, ιδιότητα μέλους. Λοιπόν, όταν θέλετε να μπει η Αλβανία, ε, θα πρέπει και η Αλβανία να το καταλάβει το μήνυμα και να εργαστεί προς την κατεύθυνση αυτή. Και βεβαίως τους είδα πολύ πρόθυμους να τα καταλάβουν. Δηλαδή, ας μην είμαστε υπερβολικά νοχελικοί και μαλθακοί, να τους λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. πολιτική κατάσταση Βεβαίω είναι αυτή που είναι, δεν θέλει η αξιωματική αντιπολίτευση να συμμετέχει στο κοινοβούλιο, είναι σοβαρό πρόβλημα αυτό. Πώ να το πω, για την αηφορία και τη βιωσιμότητα του δημοκρατικού συστήματος και την προστασία του. Και ειλικρινά ε, πιστεύω, ελπίζω να ε, αλλάξει κάτι η επίσκεψη στο Κοινοβούλιο. Κάτι άλλο τώρα εργαζόμενοι προς την κατεύθυνση απελευθέρωσης βίζας, μας βοηθάει. Βελτιώνεται και η επίδοση της χώρας στην καταπολέμηση του τράφικινγκ και του οργανωμένου εγκλήματος. Βεβαίως δεν τα έχουν καταφέρει ακόμα και θα πρέπει και αυτό να το λέμε ότι χρειάζονται και άλλες προσπάθειες για να βελτιωθεί η κατάσταση. Ε, καλό να του συγχαίρουμε. Και για τα θέματα της προστασίας του περιβάλλοντος και την πυρηνική ενέργεια. Και βέβαια δεν μπορεί να υπαγορεύσεις σε μια υποψήφια χώρα ή σε μια ενδεχομένω υποψήφια ή σε ένα κράτος μέλος τι θα κάνει, δεν θα κάνει. Αλλά εγώ συμφωνώ με τον εισηγητή ότι η πυρηνική ενέργεια δεν είναι αηφόρο, δεν είναι ανανεώσιμη, πηγή ενέργειας και βεβαίως παραμένει πολύ επικίνδυνη. Αν μη τι άλλο, εγώ δεν θα τους διαφήμιζα, δεν θα προωθούσα τέτοιες μορφές ενέργειας, παρά μόνο αηφόρες μορφές και ανανεώσιμες. Οι πράσινοι λοιπόν θα κάνουν τροπολογίες προς την κατεύθυνση αυτή και για την πυρηνική ενέργεια. Αυτά προς το παρόν, Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Thank you very much. Uh, Mr. please. Ευχαριστώ κύριος Μάτλεν. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ ε, τον εισηγητή για την έκθεσή του. Όπως είπε ήδη η κυρία Σαρχεντίνη, νομίζω ότι είναι θετική η έκθεση και τα βλέπετε ρόδινα. Έχετε βάλει κόκκινα γυαλιά ή ρόδινα γυαλιά και τα βλέπετε όλα ρόδινα. Ας πούμε, διαφθορά χρειάστηκε ε, είδατε στη Βουλγαρία και στη Ρουμανία πόσα χρόνια για να γίνουν κάποια βήματα. Δεν έχω την εντύπωση ότι είναι εύκολο να βγει κανείς από μια νοοτροπία, από μια κουλτούρα που επικρατεί. Δεν είναι καθόλου εύκολο. Και τώρα του πούμε μπράβο, συγχαρητήρια, τι καλά που τα κάνατε. Όχι, νομίζω ότι αυτό είναι εκτό τόπου και χρόνου, γιατί το έχουμε δει και σε άλλε χώρε που υπάρχει μεγάλη διαφθορά ή υπήρχε. Να δούμε τι επιδόσει τη Αλβανία λοιπόν. Τι διαπιστώνουμε. Βουλγαρία και Ρουμανία ε, είναι καλύτερα από την Αλβανία. Ε, είναι στη θέση 71 η Αλβανία και ακόμα και η Κολομβία και η Ρουάντα είναι σε καλύτερη μοίρα για τη διαφθορά. Ε, η οποία Αλβανία, κυρίες και κύριοι, είναι στη θέση 95. 71 είναι η Βουλγαρία, η Ρουμανία, επόμενες που σας είπατε γύρω στην 89 ε, και 95 Αλβανία. Τι να τη πούμε, μπράβο σα και συγχαρητήρια που καταπολεμάτε τη διαφθορά. Είναι ένα γενέ τμήμα της κουλτούρας, της νοοτροπίας εκεί πέρα και θα πρέπει να το τονίσουμε ότι εκεί πραγματικά χρειάζονται μεγάλες αλλαγές. Αλλιώς θα βάλουμε πάλι και άλλη χώρα που δεν θα έχει καταπολεμήσει τη διαφθορά. Ό, τα ίδια είδαμε και με τη Ρουμανία και τη Βουλγαρία και θα μπει και η Κροατία. Και αυτό είναι ο στόχος τελικά, το είπε και η κυρία Σαρχεντίνη. Ε, και είναι κακό να ενθαρρύνεις κάποιον που έχει τέτοια επίπεδα διαφθοράς και να τα ωρεοποιείς. Και κάτι άλλο πάλι, ε, θέμα νοοτροπίες. Από το 92 είναι μέλος της Ισλαμικής Διάσκεψης η Αλβανία. Και ε, στη διάσκεψη αυτή ε, περιορίζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα, τα δικαιώματα του παιδιού και θέλουν τη σαρία τα μέλη της Ισλαμικής διάσκεψης. Μα αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα μεταξύ των Ισλαμικών κρατών. Και σε μεγάλο βαθμό είναι μουσουλμανική χώρα η Αλβανία και επαναλαμβάνω είναι μέλος της διάσκεψης Ισλαμικών κρατών. Και αυτό ε, έρχεται σε, κατάφορη ε, παραβίαση των όσων πρεσβεύουμε εμείς στην Ευρώπη. Και πώς θα γίνει ένα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης να είναι και μέλος της Ισλαμικής Διάσκεψης. Δεν υπάρχουν αυτά τα πράγματα. Και θέλω να ρωτήσω τον εισηγητή ε, τι λέει γι' αυτό, λίγο να το κοιτάξει, τι έχει συζητήσει εκεί, τι επαφές έχει για τη Σαρία. Να το μελετήσετε αυτό το θέμα παρακαλώ. Και δεν νομίζω ότι μπορεί ένα κράτος να είναι μέλος της Ένωσης και ταυτόχρονα μέλος της Ισλαμικής Διάσκεψης. Παρακαλώ κοιτάξτε το ως Ρουμάνος κανονικά ε, θα έπαιρνα στον πειρασμό να σας απαντήσω, αλλά επειδή είμαι πρόεδρος, δεν σας απαντώ. Κύριος Αλαβράκος. Κύριε Πρόεδρε, όσο προχωράω στην οικία, προσπαθώ να ισορροπήσω μεταξύ της επίοικιας και του ρεαλισμού. Όλες οι εκθέσεις που έρχονται εδώ για υποψήφιες χώρες προερχόμενες από τα τέως ανατολικά κράτη διαπνέονται από ένα πνεύμα επίοικιας, το οποίο θέλω να προσχωρήσω διότι πιστεύω ότι κάθε άνθρωπος και κάθε χώρα έχουν ένα δικαίωμα στη ζωή και ένα δικαίωμα να έρθουν κοντά στον ήλιο, τον ήλιο αυτόν που όλους μαζί. Όμως, ο ρεαλισμός μας τι λέει για την Αλβανία. Είναι μια χώρα που δεν έχει οικονομία. Είναι μια χώρα που έχει μια ανεργία γύρω στο 33%. Είναι μια χώρα που έχει άμορφη ε, ε, προσαρμογή σε ένα οικονομικό στάτους ή σε ένα οικονομικό μοντέλο. Παράλληλα όμως δεν πρέπει να παραγνωρίζει κανείς ότι η Αλβανία είναι μια χώρα των Βαλκανίων. Και επειδή είπατε ότι είστε κι εσείς Ρουμάνος, ξέρετε πολύ καλά ότι τα Βαλκάνια είναι ο φτωχός νότος. Τα φτωχότερα κράτη του νότου. Κάποτε η Ρουμανία, από την οποία κατάγεστε, ήταν ο στοβολώνας της Ευρώπης, όπως ξέρετε. Τώρα δεν είναι. Τώρα έχει προβλήματα. Τώρα έχει προβλήματα η ίδια η Ελλάδα, η οποία έχει, ήταν η καλύτερη χώρα μέσα στα Βαλκάνια. Ήταν η μόνη χώρα του δυτικού κόσμου στα Βαλκάνια, όπως ξέρετε, η μόνη χώρα η οποία είχε κοινοβούλιο από το 1844. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι προσπαθούν να έχουν ένα κοινοβούλιο από το 90 και μετά. Άρα εδώ έρχεται το θέμα επίοικειας. Πρέπει να δούμε ότι οι άνθρωποι αυτοί πρέπει να βοηθηθούν τις ταλαιπωρίες που ζήσαν στο παρελθόν και ιδιαίτερα η Αλβανία η οποία ήταν η πιο σκληρή ε, χώρα στην περιοχή των ε, Βαλκανίων και είχε βασανιστεί από το καθεστώς Χότζερ και πρέπει να ζήσει σε κάποια στιγμή και να απολαύσει ορισμένα αγαθά που προσφέρει αυτή τη στιγμή ο σύγχρονος κόσμος. Όμως δεν πρέπει να παραβλέπουμε το εξής πρέπει να μας προβληματίσει και να καταλάβουμε τώρα πια τι ρόλο έχει παίξει η Ελλάδα. Η Αλβανία, η έκθεση για την Αλβανία είναι ένα θέμα προβληματισμού όλων των συναδέλφων για το τι ρόλο έχει παίξει η Ελλάδα στην περιοχή. Η Ελλάδα που κράτησε τη Δύση στην περιοχή, η Ελλάδα που κράτησε τη Δημοκρατία στην περιοχή, η Ελλάδα που κράτησε και κρατάει αυτή τη χώρα από πλευράς επενδύσεων. Και η Ελλάδα η οποία αυτή τη στιγμή έχει μια εκτεράστια οικονομική ταλαιπωρία η οποία εν πολλής οφείλεται στη βοήθεια των γειτονικών της κρατών χωρίς την βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έπρεπε να έχει. Σταματώ εδώ κύριε Πρόεδρε, φαντάζομαι ότι συμφωνείτε, το χαμόγελό σας είναι, δείχνει ότι συμφωνείτε μαζί μου, αλλά παρακαλώ και οι συνάδελφοι να καταλάβουν τι ρόλο έχει παίξει η Ελλάδα στα Βαλκάνια. Ευχαριστώ. Uh, Τον εαυτό μου προσπαθώ να συμφωνήσω. Καταλαβαίνω πάντως θέλετε να πείτε. Ο κύριος Χατζηγεωργίου έχει το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, νομίζω ότι είναι καλό να ξεκινήσουμε από μια από ειλικρινή συγχαρητήρια για τη δουλειά του συναδελφού. Το λέω αυτό όχι γιατί συνήθως αυτό είναι που κάνουμε όταν ξεκινούμε μια συζήτηση επί ενός ζητήματος που υπάρχει ένας ραπορτέρ, αλλά γιατί νομίζω ότι έχουμε μπροστά μας μια ανάλυση που προέρχεται από έναν άνθρωπο της περιοχής, θέλω να το τονίσω αυτό, που γνωρίζει τα πράγματα και που η ανάλυση που έκαμε με τις επαφές που έκανε στην Ελβανία μας έδωσε αυτό το σημαντικό αποτέλεσμα. Μένω λίγο στο γεγονός ότι είναι καλό να ξέρει κανείς αυτού του τύπου τις χώρες και την ιστορία τους και την γεωγραφία τους και τα προβλήματά τους, γιατί έχω ακούσει συναδέλφους που λένε «Μα έχει προχωρήσει η δημοκρατία της ε, Αλβανίας». Ασφαλώς και έχει προχωρήσει, αλλά το να λέμε ότι λειτουργεί παρότι δεν πάει η αντιπολίτευση και ψηφίστηκαν 150 νόμοι, είναι μια σχετική υπερβολή. Και αν θέλει κάποιος να βοηθήσει πρέπει να δει το πρόβλημα να το κρατήσει στο μέγεθός του, να μην το μικράνει, να μην το μεγαλώσει. Και αυτό είναι που κάνει το, το, η συγκεκριμένη ανάλυση που έχουμε μπροστά μας από τον συνάδελφο τον κύριο Χουντή. Κρατάει τα πράγματα στο μέγεθος τους. Να μην τρέξουμε προς μια κατεύθυνση η οποία στο τέλος μπορεί να βλάψει τον οποιοδήποτε στόχο. Είπε ο συνάδελφος ο κύριος Χουντής να μην παρέμβομαι με δηλώσεις τέτοιες που θα προκαλέσουν παραπάνω πολιτικές εντάσεις και συγκρούσεις στην περιοχή. Ε, όποιος ξέρει όχι μόνο την Αλβανία και άλλες χώρες της περιοχής και πιο κάτω προς τον νότο και λίγο πιο πάνω ξέρει ότι οι διατυπώσεις που προέρχονται από δημοκρατίες του τύπου που ξέρουμε στη Δύση ε, προκαλούν μια ενόχληση. Αξιοποιούνται ή χρησιμοποιούνται πολλές φορές με ένα τέτοιο τρόπο που σίγουρα δεν υποβοηθεί προς την κατεύθυνση ε, τις σκέψεις που έχουν αυτοί που τις, ε, ε, καταθέτουν. Μια κουβέντα για, για την πυρηνική ενέργεια. Συμφωνώ με την συνάδελφο από τους Πράσινους και τον συνάδελφο τον κύριο Χουντή. Δεν είναι η πυρηνική ενέργεια μια ανανεώσιμη πηγή ενέργειας εμπεριέχει πολύ σοβαρούς κινδύνους για την ανθρωπότητα, μακάρι να μην τους δούμε ποτέ μας. Μιλώ για την ενέργεια που παράγεται για ειρηνικούς σκοπούς, γιατί για την άλλη νομίζω ότι δεν έχουν πολύ πολλές αμφιβολίες. Είναι μια διαδικασία η οποία εμπεριέχει πάρα πολύ σοβαρούς κινδύνους και νομίζω ότι πρέπει η ανθρωπότητα και η Ευρώπη να δείξει το δρόμο προς αυτή την κατεύθυνση της μείωσης και της εξάλληψης, αν είναι δυνατόν, της ενασχόλησής μας με αυτό το, το είδος της ενέργειας, πολύ περισσότερο μάλιστα να το ονομάζουμε και ε, ανανεώσιμη πηγή ενέργειας. Γι' αυτό εγώ παρακαλώ κλείνω με αυτό τους συναδέρφους που είχαν έτσι πολύ έντονη άποψη ε, απέναντι στην ανάλυση που έχουμε μπροστά μας, να κατανοήσουν ότι οι δικές τους τοποθετήσεις δεν πηγαίνουν προς την κατεύθυνση που ήδη έχουν βάλει σαν στόχο. Ευχαριστώ. Uh, Ευχαριστώ. Ο κ. Πιέρ Μιρέλ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καταρχάς, να ευχαριστήσω τον κύριο Χουντή για την πολύ καλή του έκθεση. Συμφωνούμε μαζί του με τις απόψεις του όσον αφορά την κατάσταση στην Αλβανία υφιστάμενη, το υφιστάμενο πολιτικό διέξοδο σαφώς εμποδίζει την διεξαγωγή σημαντικών μεταρρυθμίσεων και ακόμα περισσότερο την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση της χώρας. Ένα από τα σημαντικά στοιχεία για την ε, πλήρωση των κριτηρίων της Κοπενχάγης είναι τα, οι δημοκρατικοί θεσμοί να λειτουργούν αποτελεσματικά και κάτι τέτοιο δεν συμβαίνει στους τελευταίους εννέα μήνες στην Αλβανία που το κοινοβούλιο δεν λειτουργεί. Και σαφώς θα πρέπει αυτό να το λάβουμε υπόψη μας όταν προτιμάσουμε τη δική μας τη γνωμοδότηση για την αίτηση προσχώρηση της Αλβανίας. Έχει περάσει το μήνυμα αυτό στους πολιτικούς ηγέτες της Αλβανίας ήδη από το Μάρτιο μέσω του Επιτρόπου Φίλε. Και αυτό το έχουμε διδαχθεί και από προηγούμενες αιτήσει για προσχώρηση από άλλες χώρες. Αν δεν υπάρχει μια σημαντική πολιτική συνένεση σε μια υποψήφια ή δυνάμει υποψήφια χώρα, τότε δεν μπορεί η δυναμη υποψηφια χωρα τοτε δεν αυτή να προχωρήσει με σημαντικές αποφάσεις, με σημαντικά μέτρα, όσον αφορά την ευρωπαϊκή της ολοκλήρωση. Τα πράγματα ουσιαστικά περιπλέκονται. Το μήνυμα λοιπόν τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή προ την Αλβανία είναι ξεκάθαρο. Καταρχά, πρέπει να λάβει χώρα στο Κοινοβούλιο ένας δημοκρατικός διάλογος, στο Κοινοβούλιο και όχι στους δρόμους. Συμφωνούμε με την κυρία Πακ ως προ αυτό. Και δεύτερον, μετά από εννέα μήνε με ένα κοινοβούλιο που δεν λειτουργεί, τόσο πλειοψηφία όσο και η αντιπολίτευση θα πρέπει να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να βρεθεί μία λύση για να καταφέρουν να επιστρέψουν σε ένα επικοδομητικό πολιτικό διάλογο. Και προκειμένου να βοηθήσουμε την Αλβανία για να βρεθεί μια λύση, είναι από τη μια υπάρχει ένας σεβασμός προς το Σύνταγμα, και από την άλλη να υπάρχει το απαραίτητο επίπεδο διαφάνειας. Μετά τις τελευταίες εκλογές, η Επιτροπή Επιτήρησης του ΑΣΕ υπέβαλε μια έκθεση, στην οποία είπανε ότι υπάρχουν ακόμα κάποια προβλήματα και είναι σημαντικά, σημαντικό να επιληθούν γρήγορα τους επόμενους μήνες τα προβλήματα αυτά. Προτού όμως γίνουν οι τοπικές εκλογές του χρόνου. Όσον αφορά τώρα τη θετική πλευρά των πραγμάτων. Όντω η χώρα έχει σημειώσει σημαντική πρόοδο όσον αφορά την ε, ελευθέρωση των θεωρήσεων, τη σχετική διαδικασία, προκειμένου να φτάσει σε απαραίτητες προδιαγραφές. Μολονότι βέβαια υπάρχουν ακόμα κάποια εκρεμή ζητήματα. Εμείς Παρουσιάσαμε χθε στην Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών τη δική μα αξιολόγηση και τη Δευτέρα στο Συμβούλιο την παρουσιάσαμε. Θα προτιμάσουμε τι επόμενε εβδομάδε και την επίσημη πρόταση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ένα σημαντικό ζήτημα το οποίο υπογράμμισε και στην εκθέση του κύριο Χουντή είναι η κατάσταση του δικαστικού συστήματο και ότι ε, πρέπει να εφαρμοστεί μια μεταρρυθμιστική στρατηγική, μια στρατηγική μεταρρυθμίσεων για το δικαστικό σύστημα. Και πάλι αυτό είναι ένα δίδαγμα, θέλετε, από προηγούμενες αιτήσεις για προσχώρηση. Είναι σημαντικότατο να μπορεί οποιοδήποτε πολίτης να προσφύγει στα δικαστήρια για να κατοχυρώσει τα δικαιώματά του και ο πολίτης και οι επιχειρήσεις. Είναι πολύ σημαντικό επίσης να λειτουργεί το σύστημα αυτό για να καταπολεμηθεί το οργανωμένο έγκλημα και είναι πολύ σημαντικό που σας είπα για το οργανωμένο έγκλημα και τη διαφθορά για την πάταξή τους. Πέρα από το ζήτημα των θεωρήσεων και την απελευθέρωση των θεωρήσεων, αυτό που μας ενδιαφέρει να δούμε και κέρις πλέον μεταρρυθμίσεις στο δικαστικό σύστημα. Και θέλουμε επίσης να δούμε και ποια θα είναι τα απτά αποτελέσματα μετά τις μεταρρυθμίσεις αυτές που έχουν εγκριθεί. Επίσης, μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης. Και αυτό θα πρέπει να γίνει, όπως άλλωστε λέγεται στην έκθεση. Είναι ένα ζήτημα πολύ σημαντικό για τον εξυγχρονισμό της Αλβανίας και είναι πολύ σημαντικό επίσης και για τον, την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση της Αλβανίας. Θεωρούμε επίσης ότι μέσα μας και ενημέρωση θα πρέπει να λειτουργούν ανεξάρτητα και ελεύθερα. Πολύ περισσότερα πράγματα θα πρέπει να γίνουν. Έχουμε καταδικάσει την στάση που κρατά κυβέρνηση απέντη στους δημοσιογράφους, κάποιες απειλές απέναντι στους δημοσιογράφους που ακούσαμε. Περισσότερα πράγματα πρέπει να γίνουν επίσης και για τις συνδικαλιστικές οργανώσεις που δεν μπορούν να λειτουργήσουν πλήρως όπως θα έπρεπε. Ένα από τα ζητήματα που είχε αρνητική επίπτωση για τα δικαιώματά τους ήταν ο νόμος για την εθνικοποίηση της ιδιοκτησίας τους που βέβαια θεωρήθηκε αντισταγματικός. Παρακολουθούμε λοιπόν πολύ κοντά την εξέλιξη του ζητήματος αυτού. Η κατάσταση των γυναικών και των παιδιών, η προάσπιση των δικαιωμάτων τους και αυτό πρέπει να μας απασχολήσει. Έχει σημειωθεί μια πρόοδος, αυτό πρέπει να το αναγνωρίσουμε, αλλά πρέπει να γίνουν ακόμα περισσότερα πράγματα προκειμένου να σταματήσει η ενδοκογενειακή βία, καθώς επίσης και η εμπορία γυναικών και παιδιών για λόγους σεξουαλικής εκμετάλλευσης. Μια θετική εξέλιξη είναι η νομοθεσία κατά των διακρίσεων η οποία εγκρίθηκε στα πλαίσια της ελευθέρωσης των θεωρήσεων. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για τις μειονότητες και αυτό το οποίο θα πρέπει να προσέξουμε αυτή τη στιγμή είναι πραγματικά να εφαρμοστεί στην πράξη αυτή η νομοθεσία. Όσον αφορά τώρα την οικονομική κατάσταση, ίσως να μην συμφωνήσουμε στο σημείο αυτό με τον εισηγητή, μόλον ότι προφανώς πρέπει να γίνουν διαρθρωτικές αλλαγές, αυτό είναι προφανές, η Αλβανία έχει μια, ένα πολύ μεγάλο τομέα της οικονομίας που σαστικά είναι παραοικονομία. Παρά όμως την κρίση, οι προοπτικές για τα επόμενα δύο χρόνια είναι εντυπωσιακέ. Ε, θα Θευχόμαστε ουσιαστικα ουσιαστικά κάποια κράτη-μέλη να είχαν πραγματικά τέτοιες θετικές οικονομικές προοπτικές. Συμφωνώ με τον κύριο Ρουτσέκ στο ότι πρέπει να αναγνωρίσουμε τον θετικό ρόλο τον επικοδομητικό ρόλο που διαδραματίζει η Αλβανία στην περιοχή. Ολοκληρώνω κύριε Πρόεδρε στο σημείο αυτό. Αυτά είναι τα βασικά ζητήματα που θέλησαμε εμείς να τονίσουμε. Σας ευχαριστώ. Σα Σας ευχαριστούμε πολύ. Τον λόγο έχει ο κύριος Χουντής για να απαντήσει. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους και τις συναδέλφισες που πήραν το λόγο, που μελέτησαν το κείμενο και που έκαναν παρατηρήσεις. Είναι πολύ βοηθητικές. Σπέβδω να πω ότι υπάρχουν παρατηρήσεις και συμπληρώσεις που επικαιροποιούν ορισμένες διαπιστώσεις, διατυπώσεις που δεν ήταν γνωστές όταν εγγράφεται το αρχικό σχέδιο ή δεν είχε εκτιμηθεί η αξία τους. Με αυτή την έννοια ότι παρέδωσε το ερωτηματολόγιο ότι μετέχει σε θεσμούς περιφερειακής συνεργασίας ε, είναι σωστό, ότι βοήθησε σε σχέση με τις γειτονικές χώρες η κατάργηση της θεώρησης της βίζας με άλλες χώρες. Αυτά είναι πράγματι θέματα που πρέπει να τεθούν. Τώρα, στη γενική παρατήρηση αν είναι θετική ή είναι λιγότερο θετική από προηγούμενη έκθεση παρά τα βήματα που έγιναν, θα σας έλεγα ότι όπου είναι δυνατόν πράγματι να κρατηθεί ζωντανό ένα μήνυμα να ενθαρρυνθεί η αλβανική κοινωνία να κάνουν τα απαραίτητα βήματα, θα το πάρω υπόψη μου. Όμως, όμως ε, ισχυρίζομαι ότι πίσω από σύντομες διατυπώσεις και για την οικονομία του κειμένου θα μπορούσα να σας πω ε, για αρκετή ώρα για διάφορα προβλήματα τα οποία ε, και από στοιχεία και από την επιτόπια συζήτηση και με τη βοήθεια όλων δείχνουν τις διαστάσεις των προβλημάτων και θα έλεγα όχι μόνο δεν δε θα έπρεπε να τις κρύψουμε αυτές τις διαστάσεις των προβλημάτων αλλά να κινηθούμε με δύο σκοπιμότητες, κατά τη δική μου άποψη. Το πρώτο, προς τις πολιτικές δυνάμεις της Αλβανίας, υπογραμμίζοντας ότι έχουν να λύσουν σοβαρά προβλήματα, ενδεχομένως να τους θυμίσουμε ότι πρέπει να έρθουν στο ύψος των περιστάσεων, θα έλεγε κανείς, και να δοθεί πολιτική διέξοδος για να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα. Αντί να εξοραίσουμε τα πράγματα και κλείσουμε εκεί. Και το δεύτερο, η δεύτερη διάσταση είναι σε μια σειρά από αυτά τα θέματα που ίσως μπαίνουν με σκληρό τρόπο, δεν το πιστεύω, παρόλα αυτά πιστεύω ότι μπαίνει αντικειμενικά, υπάρχουν περιθώρια και προτάσεων πώς μπορούμε να βοηθήσουμε οι άλλες γειτονικές χώρες, η Ευρωπαϊκή Ένωση συνολικά, για να αντιμετωπιστούν αυτά τα ζητήματα. Σας αναφέρω μόνο ένα θέμα που είναι η καταγραφή των παιδιών. Δεν καταγράφονται όλα τα παιδιά όσα γεννιούνται στα νοσοκομεία, άλλα δεν γεννιούνται στα νοσοκομεία και άλλα για πολλού και διαφόρου λόγου γεννιούνται σε άλλε χώρε. Και υπάρχει ένα μεγάλο κενό. Αν δεν βοηθήσουν στην προκειμένη περίπτωση και οι άλλε χώρε, στην προκειμένη περίπτωση και η χώρα μου, η Ελλάδα, προκειμένου να αντιμετωπιστεί αυτό το θέμα, καταλαβαίνετε τι προβλήματα μπορεί να δημιουργήσει στα νέα παιδιά, ε, στα παιδιά όλη αυτή η κατάσταση. Απλώ το ανέφερα σαν παράδειγμα τι βοήθεια χρειάζονται σε μια σειρά ζητήματα. Τώρα, για την πολιτική κρίση. Εδώ, αγαπητοί συνάδελφοι, υπογραμμίζω για άλλη μια φορά ότι πέρα από αυτά που λέγονται από τα δύο μεγάλα κόμματα, τα οποία κατά τη γνώμη μου έχουν την ευθύνη για το σε ποιο επίπεδο βρίσκεται το πολιτικό σύστημα, καθώς τις τελευταίες δεκαετίες εναλλάξ κυβέρνησαν ε, την Αλβανία, συζήτησα με όλα τα κοινοβουλευτικά κόμματα και σα είπα και με την κοινωνία των πολιτών. Και ορισμένε παρατηρήσει σε σχέση με τη λειτουργία του πολιτικού συστήματο, του εκλογικού συστήματο, προκύπτουν από στοιχεία καταθέσει που κάνουν όχι μόνο τα δύο μεγάλα κόμματα, επαναλαμβάνω. Και η αποφυγή να πάρουμε θέση, κατά τη δική μου άποψη, θα πρέπει να συνιστά υπεύθυνη, συνιστά υπεύθυνη στάση αντί να δούμε ανάλογα με την κομματική συγγένεια του καθενός μας, της κάθε ομάδας, προ τα που πρέπει να ρίξουν το βάρο, ότι έχει δίκιο ο κύριο Μπερίσα ή έχει δίκιο ο κύριο Ράμα. Κατά τη γνώμη μου, αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να επισημάνουμε τα προβλήματα, να επισημάνουμε στη βάση ποιων αρχών, να επισημάνουμε ότι το Κοινοβούλιο δεν λειτουργεί και πρέπει να λειτουργήσει σε κάθε περίπτωση και ότι η λύση πρέπει να προκύψει μέσα από το δικό του διάλογο, μέσα από τη δική ειναι να επισημανουμε τα προβληματα να υπεσημανουμε στη βαση ποιων αρχων να υπεσημανουμε οτι το σεβασμό του συντάγματο. Δεν μπορούμε, κατά την άποψή μου, να υποδείξουμε λύσει. Για την οικονομία, ε, είπα και εισηγητικά ότι σαφώς οι διατυπώσεις εκεί πρέπει να βελτιωθούν. Όμως να μου επιτρέψετε και μπορεί να μην γραφτεί στο κείμενο να εκφράσω τις εξής επιφυλάξεις σχετικά με το ποια είναι τα οικονομικά προβλήματα της Αλβανίας. Θέλω να θυμίσω στους συναδέλφους που έκαναν την παρατήρηση ότι η Αλβανία ή και άλλες χώρες ε, μέσα σε περίοδο κρίσης εμφανίζουν υψηλό ποσοστό, σχετικά υψηλό ποσοστό του ΑΕΠ, αύξηση, ανάπτυξη του ΑΕΠ, ότι η Ελλάδα, από την οποία προέρχομαι, που βρίσκεται τώρα στη μάτι, στο μάτι του κυκλώνα της κρίσης, για τα περισσότερα χρόνια, πριν δύο χρόνια, για μια δεκαετία ουσιαστικά είχε τους υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή ήταν μια ανάπτυξη έολη, μετέωρη, δεν στηριζόταν πουθενά και, εν πάση περιπτώσει, αποδείχθηκε ότι δεν είχε βάση. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, αυτή η πρόβλεψη να, ε, ε, ενδεχομένως αδικούσε τις προσπάθειες της Αλβανίας και εκεί να το διορθώσουμε ότι έχει κάνει βήματα κτλ. Όμως ε, θα ήθελα όσο αφορά το τι μπροστά μπορεί να βρει η αλβανική οικονομία της Αλβανίας αν δεν πάρει τα απαραίτητα μέτρα και εδώ θα το ξαναδιατυπώσω το κείμενο τι σημαίνει απαραίτητα μέτρα νομίζω ότι θα, θα εισπράξει έστω και καθυστερημένα πράγμα που δεν εύχομαι την κρίση. Τέλος, για το ενεργειακό πρόβλημα είναι πάρα πολύ κρίσιμο. Ε, επειδή ξεκινάει τώρα τον, ε, ας πούμε, τον ενεργειακό της ε, ανασυγκρότηση, νομίζω ότι η προτροπή να δοθεί προτεραιότητα στις ανανεώσιμες πηγές πρέπει να έχει κυρίαρχο ρόλο. Και το δεύτερο, σε σχέση με την πυρηνική ενέργεια, θα σας έλεγα, επειδή προέρχομαι, όπως είπα επανειλημμένα, από το χώρο των Βαλκανίων, η περιοχή είναι πολύπαθη, έχει ακόμα πηγές ένα ενδεχόμενο νέο πυρηνικό εργοστάσιο στον χώρο της Αλβανίας δεν θα ήταν καλός, καλό σημάδι για την βελτίωση των σχέσεων και για την ασφάλεια γενικά της περιοχής. Υπάρχει έντονη διάθεση, ένα κίνημα για Βαλκάνια χωρίς πυρηνικά που συγκεντρώνει ευρύτατη υποστήριξη και στο πνεύμα αυτό η υπογράμμιση νομίζω ότι θα βοηθούσε την αντιμετώπιση αυτού του θέματος Ξαναλέω, αυτή τη στιγμή από την αρχή ανασυντάσσονται ενεργειακά στον χώρο αυτό. Ε, αυτά κύριε Πρόεδρε και τις άλλες παρατηρήσεις, τις παρατηρήσεις και τις τροπολογίες θα κάνω μια προσπάθεια και με τους συναδέλφους που τις διατύπωσαν, με τους α, εισηγητές από τις άλλες ομάδες και με την κατάθεση την ημέρα των τροπολογιών να το βελτιώσω, να βελτιωθεί το κείμενο. Thank you much. After all, this is the first time Ευχαριστώ πολύ. Κοιτάξτε, δείτε, έτσι κι αλλιώς είναι μια πρώτη ανταλλαγή απόψεων για ε, την έκθεση αυτή και μέχρι τις 12 το μεσημέρι της 5ης Μαΐου έχουμε χρόνο για την κατάθεση των τροπολογιών μας. Ευχαριστώ όλους όσοι συμμετείχαν στη συζήτηση και θέλω να περάσουμε τώρα στο επόμενο θέμα που είναι και κλεισμένο των θυρών και θα παρακαλούσα όλους εκείνους ε, και ε, και των φίλων μας από το Συμβούλιο και την Επιτροπή ε, που δεν θα είναι παρόντες να επανέλθουν στη συνέχεια για το τελευταίο θέμα. Έτσι λέει η διαδικασία και θα πρέπει να τη σεβαστούμε. Δηλαδή πρώτα το κεκλεισμένο των θυρών και μετά το άλλο θέμα να ξανάρθετε.